Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα αρχίσω με λίγα λόγια στα πορτογαλικά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για μένα αποτελεί μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας στο σώμα αυτό της Δημοκρατικής Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω εδώ τις ιδέες μου και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η ιστορία μου είναι μια ευρωπαϊκή καθαρά ιστορία. Γεννήθηκα σε μια όμορφη πόλη στο νότο της Πορτογαλίας, όπου οι περισσότερες οικογένειες έζησαν υπό συνθήκες σοβαρής ένδυας. Αυτή η περιφέρεια ευεργετήθηκε κατά πολύ από την σκληρή εργασία των πολιτών αλλά και από τα μέσα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Μεγαλώνοντας είδα από πρώτο χέρι τον ε, ζωτική σημασία ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη στην ε, παγιοποίηση της νέας μας δημοκρατίας όπως ίσχυσε για την Ελλάδα και την Ισπανία. Είδα πώς η Πορτογαλία μπόρεσε να αδράξει τις ευκαιρίες ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας που μας έδωσε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ζωή μου σηματοδοτήθηκε από ε, γεωγραφική κινητικότητα και άναντι κινητικότητα που μας ε, δίδει, μπορεί να μας δώσει μόνο η Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Έτσι έγινα ο άνθρωπος, ο πολίς και ο πολιτικός που είμαι σήμερα. Από την γενέτειρά μου κινήθηκα προς την πρωτεύουσα της ε, χώρας μου εξαιτίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος που η δημοκρατία δημιούργησε χωρίς αποκλεισμούς. Οι γονείς μου είχαν ένα στόχο, να στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο και τα κατάφεραν. Αυτό που δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ήταν ότι μία ημέρα ένα από τα παιδιά τους ε, θα μετέβαινε από τη Λισαβόνα στο Παρίσι χάρη σε ένα μεγάλο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα Έρασμους. Το Έρασμους ήταν το σημείο κατακλίδα για τη ζωή μου και αυτό ισχύει όχι για μένα αλλά και για τη γενιά μου. Εγώ είμαι από τους πρώτους ε, στη χώρα μου που ευεργετήθηκα από αυτό το πρόγραμμα και θα σας πω τώρα λίγα λόγια και στα γαλλικά. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια στα γαλλικά, διότι και η Γαλλία είναι κατά κάποιο τρόπο η χώρα μου. Στη Γαλλία τελείωσα τις σπουδές μου και στην Γαλλία άρχισα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία ως μηχανικός. Στη Γαλλία γνώρισα τη γυναίκα μου και στη ε, Γαλλία επίσης παντρεύτηκα στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού. Μετά μεταβήκαμε στις ΗΠΑ όπου συνέχισα τις μελέτες μου και τις σπουδέ μου και είδα ποια είναι η προοπτική του να είναι κανείς Ευρωπαίος. Μπορεί κανείς να δει πιο καθαρά τις ε, μοναδικές ευρωπαϊκές αξίες και τον πολιτισμό τον οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε για τα παιδιά μας. Μετά από τη Βοστόνη πήγα στο Λονδίνο όπου γεννήθηκαν δύο από τα τρία μου παιδιά και έζησα για τέσσερα χρόνια εκεί σε μία από τις πιο ζωντανές και εκπληκτικές πόλεις του κόσμου. Μετά επέστρεψα στην Πορτογαλία όπου ε, ασχολήθηκα με επιχειρήσεις. Ήμουνα διευθυντικό στέλεχος και δημιούργησα και τη δική μου επιχείρηση. Το 2011 εξελέγεν βουλευτής και διορίστηκα από την κυβέρνηση ως υπουργός και μπόρεσα να δω ποια ήταν η κατάσταση της Πορτογαλίας σε μια στιγμή εθνικής και ευρωπαϊκής κρίσης. Η ιστορία μου είναι μια ευρωπαϊκή ιστορία. Τώρα ενώπιόν σας θέλω να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο έτσι ώστε να μπορέσω να υπηρετήσω την Ευρώπη και να της δώσω και εγώ αυτό, αυτά που μου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια δεσμεύομαι να συνεργαστώ μαζί σας για την ε, στεναρή πρόοδο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, όπως ξέρετε, ο οριστής Ζαν ε, Κλοντ ε, Juncker μου ανέθεσε τον τομέα της έρευνας επιστήμης και καινοτομίας. Αναλαμβάνω αυτή την πρόκληση με μεγάλο ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση, διότι πιστεύω στην πολιτική ατζέντα του οριστέντος Προέδου, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ε, εργασία στην Ευρώπη μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας και της αριστείας, την έρευνα και την επιστήμη. Η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να προωθήσω τις συνθήκες πλαίσιο που θα επιτρέψουν την ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία να προχωρήσουν. Θα καταφέρναμε πολλά, πολύ περισσότερα αν είχαμε λιγότερα προσκόμματα και αν είχαμε μία αναπτυξιακή ικανότητα να προσελκύσουμε παγκοσμίως ταλέντα. Επίσης, αυτό αφορά, την πεμπτουσία της, αυτό αφορά και την πεμπτουσία της καινοτομίας. Για να προωθήσουμε τις συνθήκες πλαίσιο θα πρέπει να δώσουμε τελική μορφή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στην Ένωση καινοτομία. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός και εποπτεία και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να προωθήσουμε συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία καθώς και τα επενδυτικά ταμεία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να προωθήσουμε τις ικανότητες και την καινοτομία. Επίσης, θα ε, επαγρυπνώ ως προς την τήρηση της διάστασης και τη συμμετοχή των δύο φύλων, διότι θεωρώ ότι το ταλέντο αφορά και τα δύο φύλλα. Η δεύτερη μου προτεραιότητα είναι να υπάρξουν αποτελέσματα ως προς τον ορίζοντα 2020. Σήμερα έχουμε, βρισκόμαστε εδώ γιατί ε, γευθήκαμε τα προνόμια τα οποία μας έδωσε μεταξύ άλλων το Κοινοβούλιο μέσα στην απέραντη σοφία του. Θα πρέπει λοιπόν τα 80 δις του ορίζοντα 2020 να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσουμε με την ατζέντα πλούστευσης όπου καταφέραμε ήδη πολλά επειδή η Επίτροπος Γκέγκαν Κουίν ήταν πολύ αποτελεσματική και με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Έτσι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέα στοιχεία στην έρευνα και την επιστήμη για να φέρουμε αποτελέσματα στον ορίζοντα 2020 θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας εφαρμόζοντας το πακέτο καινοτομίας και επενδύσεων, προωθώντας τα, μέσα, τα χρηματοδοτικά μέσα καινοτομίας, περιλαμβάνοντας τις ΜΜΕ και εστιάζοντας την προσοχή μας στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην ε, χαμηλή χρήση του άνθραγα καθώς και των ανανεώσιμων. Πιστεύω ότι οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να προωθήσει τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις υπό την αιγίδα του οριστέντος Προέδρου Γιούνκερ. Η τρίτη μου προτεραιότητα θα είναι να υποστηρίξω την αριστεία στην ε, έρευνα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την δημιουργική ελευθερία που διέπει την εργασία των ερευνητών και των επιστημόνων. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σχέδια σε δύσκολους τομείς. Πιστεύω ότι έτσι αυτό το ριάκι θα οδηγήσει στα βαθιά ποτάμια της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Γι' αυτό και υποστηρίζω το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Επίσης θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε μια νέα γενεά νέων ταλαντούχων και δυναμικών ερευνητών. Μέσα στα πλαίσια αυτών των τριών προτεραιοτήτων θα πρέπει να επιταχύνουμε το βήμα μας για να ακολουθήσουμε τη, τις παγκόσμιες εξελίξεις μέσα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, προσμένω τις ερωτήσεις σας σήμερα και αν διοριστώ μέλος της Επιτροπής Πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία τα επόμενα έτη. Όταν υπηρέτησα την εθνική κυβέρνηση, εργαζόμουν κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή για να άρω τα προσκόμματα, να απλουστεύσω τις διαδικασίες και να δημιουργήσω νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους. Εάν ε, οριστώ επίτροπος, θα ακολουθήσω την ίδια αυτή όθηση, διότι πιστεύω στη δύναμη της έρευνας, της επιστήμης και της καινοτομίας. Θα εστιάσω την προσοχή μου στα αποτελέσματα, στα καθαρά αποτελέσματα. Στην ευρωπαϊκή μου ιστορία και με βάση την πολιτική μου πείρα εργάστηκα μέσα σε θεσμικά πλαίσια και σε διάφορους τομείς. Ε, προσπάθησα να αποτρέψω τα στέγανα, τα τεχνητά στέγανα, διότι πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εργαστεί συνεργατικά. Θα πρέπει λοιπόν, εάν διοριστώ, να υπηρετήσω την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, διότι αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ε, βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρώπη και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε και τώρα θα περάσουμε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων από πλευρά ε, των πολιτικών ομάδων. Θα ακούσουμε τους ομιλητές. Ο κύριος Κρίστιαν Έλερ από πλευράς του ΕΛΚ. Καλώς ορίσατε κύριε Μέδας και καλώς ορίσατε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτη μου ερώτηση θα ήταν η εξή. Ε, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα προέκυπτε μία αύξηση της αποδοτικότητας τα επόμενα χρόνια μέχρι τα 11 δισεκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική ατζέντα. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά προσκόμματα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και ποιε είναι οι προτεραιότητέ σα για να πετύχετε του στόχου σα, τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών, καθαρά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να απαντήσουμε να ακούσουμε την απάντησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Έιλερ για την ερώτηση που μου κάνατε. Δήλωσα και πιστεύω απόλυτα ότι ο ευρωπαϊκός χώρος ε, έρευνας είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρώπη. Όχι μόνο επειδή Πρόκειται για την, ένα έργο για την έρευνα, την κοινοτομία και την επιστήμη, αλλά γιατί είναι σημαντικό για όλο το ευρωπαϊκό οικοτόμημα. Ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας έχει ως στόχο να άρει τα εμπόδια, τα προσκόμματα, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη συνεργασία, καλύτερη ροή πληροφοριών. Αλλά, για να απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας, θεωρώ ότι τα πιο πολλά εργαλεία που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη υπάρχουν. Αυτό που λείπει τώρα είναι το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό με τα, κράτα, με τα κράτη-μέλη. Πώς θα εφαρμοστούν από πλευράς κρατών μελών τα εργαλεία αυτά. Και θα ήθελα να τονίσω τρία πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην παρούσα φάση. Το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε καλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των εθνικών σχεδίων ανάπτυξης και έρευνας. Γιατί? Για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό, την αλληλεπικάλυψη. Κατά δεύτερον, υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που αφορά την έλλειψη διαφάνειας, που εξακολουθεί σε κάποιες περιπτώσεις να υφίσταται σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και κατά τρίτον, να συνεχιστεί η προώθηση της διάστασης του φίλου και να καταπολεμηθεί η ανισότητα μεταξύ των φίλων που είναι κάτι πραγματικά αδίκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, το 2015 καταστράφηκε ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα είναι πραγματικά αναλέητος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Κάρλος Ζωρίνιο από σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Θα ήθελα να χαιρετήσω ε, τον υποψήφιο επίτροπο και να τον καλωσορίσω στην αρχή σας παρουσίαση επιδείξατε μια ε, τολική ε, συμμόρφωση με το πρόγραμμα του Jean-Claude Juncker. 300 εκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν ε, για να τονωθεί η οικονομία της Ευρώπης μέσα από διάφορα τεχνολογικά σχέδια. Ταυτόχρονα όμως ε, θέλει η Ευρώπη να περικόψει τα κονδύλια του ορίζοντα 2020. Είναι απαραίτητο αυτό, αλλιώς δεν έχει αξιοπιστία το πρόγραμμα του Ζαν κλοντ Juncker. Τρεις ερωτήσεις έχω. Τι πιστεύετε, μπορείτε να πείσετε το Συμβούλιο όχι μόνο να μην περικόψει τα κονδύλια αλλά και να ενισχύσει το πρόγραμμα ορίζοντας 2020. Δεύτερον, ποιο ποσοστό του προγραμμου jean Jean-Claude Juncker θα μπορέσετε να διοχετεύσετε στην έρευνα, επιστήμη και καινοτομία. Και τρίτον, ποια είναι η στρατηγική σας ε, για να ε, συνδεθεί ο ορίζοντας 2020 με το πρόγραμμα πράσινης και θα, ε, ε γαλάζιας ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε Βουλευτά για τις ερωτήσεις σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσω και πορτογαλικά και να σας χαιρετήσω και ε, ε προσωπικά. Τα 300 δις ε, που ανέφερε ο Ζαν Κλοντ και θα επιβεβαιωθούν από τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν είναι ένα πακέτο πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Εάν εγκριθεί η υποψηφιότητά μου, αυτός ακριβώς θα είναι ο στόχος μου. Θα προσπαθήσω να δείξω την θεμελιώδη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τη μελλοντική ανάπτυξη. 62% της ανάπτυξης προήλθε από την καινοτομία κατά την περίοδο 1995 έως 2007. Γι' αυτό στο νέο πακέτο 300 δις θα είναι βασικός πυλώνας η έρευνα και η καινοτομία και εγώ θα υπερασπιστώ αυτή την αρχή. Θα ήθελα επίσης να σας πω πως όταν ε, κοιτάζουμε το μέλλον προσπαθούμε ως Ευρωπαίοι να συνειδητοποιήσουμε την σημασία αυτού του τομέα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το έχουμε συζητήσει στην αλληλογραφία μας, το 2009-2010 θα θυμάστε αυτά που είχαμε συζητήσει η διαλογραφία στην Πορτογαλία Ε, σας ε, μετέφερα ένα μήνυμα υπέρ της καινοτομίας και της ανάπτυξης και δεν έχει αλλάξει αυτή μου η πεποίθηση. Αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσω και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Hans Olaf Henkel από πλευράς του ECR. Κύριε Μετάσα, σας μιλώ από τα μετόπισθεν. Ελπίζω να μην το πάρετε προσωπικά αυτό. Μας ε, παρουσιάσατε τις προτεραιότητές σας, ε, όλες ε, σωστές. Ωστόσο, κάτι μου λείπει. Ακόμα και αν κάναμε όλα όσα σκοπεύουμε να κάνουμε στην Ευρώπη, αυτό θα καλύψει μόνο το 6% των, συνολικών δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη. 94% δηλαδή είναι στα χέρια των κρατών μελών. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Τι κάνατε για να διασφαλίσετε ότι οι χώρες επιτέλους θα δαπανίσουν τα χρήματα αυτά για την έρευνα και την ανάπτυξη. Το έχουν υποσχεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό άλλωστε. Αλλά μόνο λίγες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που το κάνουν. Η Ελβετία προφανώς, η Σουηδία, η Φιλανδία. Ε, πιστεύετε ότι χρειάζεται μία επιπλέον προτεραιότητα προκειμένου να πιστούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κάνουν ό,τι έχουν υποσχεθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας, αλλά νομίζω ότι αναφερθήκατε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο βρίσκεται άλλωστε και στην καρδιά του χαρτοφυλακίου αυτού. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, πώς μπορούμε να διαβιβάσουμε το μήνυμα του πόσο κρίσιμη σημασίας είναι η έρευνα, η επιστήμη και η κοινοτομία αναφέρθηκα σε αυτούς τους εντυπωσιακού ε, στα εντυπωσιακά ποσοστά ότι το 62% της ανάπτυξης της Ευρώπης στις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται στην έρευνα, την επιστήμη και την ανάπτυξη. Κοιτώντας λοιπόν τα προγράμματα που έχουμε στο χαρτοφαγγλάκιο ορίζοντας 2020, θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους μόχλευσης μεταξύ των προγραμμάτων, όπως τα αντιθετικά ταμεία, που για την καινοτομία έχουν μεγάλη συμμετοχή, μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να εναρμονιστούν ε, τα σχέδια δράσης μεταξύ των κρατών μελών. Έχουμε προγράμματα και υποδομές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλη την Ένωση. Γιατί αν υπάρχει μια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η επιστήμη, η έρευνα και η ανάπτυξη και η καινοτομία. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στις χώρες αυτές πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω ότι ο ρόλος του χαρτοφυλακίου αυτού θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερος, ακόμα πιο έντονος σε ό,τι αφορά και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό υφίσταται μεν ως στοιχείο, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να τονιστεί περαιτέρω. Ευχαριστώ.